Voilà, allez. Ναι. Bonjour à tous. Dans le cadre des discussions sur le cluster 1 de cette audition, intitulée Le trafic. Έχουμε να μιλήσουμε για το, εμπόριο, το παράνομο εμπόριο όπλων. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάρσε, που είναι υπεύθυνο για σοβαρή εγκληματικότητα της Ευρωπολίτη, κυρία Σέντερα από την ομάδα ΣΟΚΤΑ που θα μας μιλήσει για παράνομο εμπόριο όπλων και για οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη βλέπω. Φάμπιο Μαρίνη, που είναι επικεφαλής του τομέα αγώνα κατά της ε, κυκλοφορίας όπλων ε, στην, Γενική, στην Κομισιόν θα μας μιλήσει για την ε, εγκληματική χρήση των όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Κομέλη, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Οπλουργών της Γαλλίας και θα μιλήσει για την, ε, ε, το παράνομο εμπόριο των όπλων. Θα έχουμε δεκάλεπτη παρουσίαση του κύριου Χόφενμπακ και δεκάλεπτη παρουσίαση του κυρίου Μαρίνη και στη συνέχεια ο κύριος Κιγκολέτη. Έπειτα θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους ε, βουλευτές που θα έχουν ζητήσει το λόγο, με προτεραιότητα για τον εισηγητή κύριο Γιακολίνο και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, ελπίζοντας πως θα καταφθάσουν που να είναι. Και όλοι καλείστε να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας σε τρία λεπτά. Έπειτα θα έχουμε τις απαντήσεις του κυρίου Μαρίνη και του κυρίου Γκολέτη. Κύριε Όφερμα, σας δίνω το λόγο. Thank you very Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα, εξ ονόματο τη ε, Europol, θα ήθελα να σα εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου. Όταν μιλάμε λοιπόν για την ε, Europol και τη γνώση που έχει για το λαθρεμπόριο όπλων και το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε δύο βασικές πηγές πληροφοριών από τα κράτη-μέλη. Το ένα αφορά τη βασική μας δουλειά που είναι η στήριξη των διασυνοριακών έρευνών για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Επιχειρησιακές πληροφορίε που λαμβάνουμε κάθε μέρα μαζί με αιτήματα στήριξης τα οποία στηρίζουμε κυρίως βεβαίως μέσω συντονισμού και ανάλυσης αυτά κάνουμε στο επίπεδο της Europol. Βεβαίως δεν χρησιμοποιούμε μόνο αυτές τις ε, πληροφορίες για να στηρίξουμε τις επιχειρησιακές ε, δυνατότητες των κρατών μελών, αλλά βλέπουμε και τις πληροφορίες αυτές με τρόπο στρατηγικό για να εντοπίσουμε εξελίξεις και μελλοντικές απειλές για να είμαστε έτοιμοι και να προειδοποιήσουμε τα κράτη-μέλη και τις διοπτικές αρχές αναλόγως. Λαμβάνουμε λοιπόν και στρατηγικές πληροφορίες. Οι πιο σημαντικές συνεισφορές αφορούν την εκτίμηση κινδύνου για σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Η αξιολόγηση αυτή του κινδύνου είναι σε μια ετήσια βάση και μπορεί να θεωρηθεί νομίζω ως μία από τις σοβαρότερες και πιο λεπτομερείς μελέτες του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζεται σε συνεισφορές των διοκτικών αρχών των κρατών μελών, αλλά και από τρίτες χώρες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες όπως η Frontex και η Eurojust και οργανισμοί όπως η Interpol και λοιποί. Επίσης, λαμβάνουμε πληροφορίες από τον ιδιωτικό τομέα και τα πανεπιστήμια όπου έχουμε οργανώσει συγκεκριμένα εργαστήρια για να είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Η μεθοδολογία έχει συμφωνηθεί από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και προβλέπει πως τα κράτη-μέλη συμπληρώνουν κάποιο ερωτηματολόγιο και τους έχουμε ζητήσει επίσης να δίνουν πληροφορίες όσον αφορά την απειλή του λαθρεμπορίου όπλων όμως. Με βάση τις αναφορές αυτές που δίνουν τα κράτη-μέλη, η απειλή από το λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων ε, είναι περιορισμένη. Μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν αναφέρει λαθρεμπόριο όπλων ως υψηλή απειλή η οποία ήταν περιορισμένη σε σχέση με άλλες απειλές του οργανωμένου εγκλήματος λόγω των ε, συνεισφορών που είχαμε από άλλα κράτη-μέλη που σχετίζονται με σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Οι ομάδες ε, που έχουμε εντοπίσει ότι εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο αυτό δεν εμπλέκονταν αποκλειστικά σε αυτό το λαθρεμπόριο. Um, all the groups Καμία, ομάδα δεν το έκανε αυτό αποκλειστικά. Ήταν λεγόμενες πολυεγκληματικές ομάδες. Ε, όπως εντοπίσαμε και στην αξιολόγηση κινδύνου, την οποία εκδώσαμε πριν από λίγες εβδομάδες. Οπότε βλέπουμε πολυεγκληματικές ομάδες που παραδίδουν τα όπλα όταν τους το ζητήσουν άλλες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος ή τα χρησιμοποιούν οι ίδιες. Φαίνεται πως το λαθρεμπόριο όπλων δεν είναι η βασική πηγή εισοδήματος. Είναι μάλλον κάτι το συμπληρωματικό που σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες. Περισσότερες δηλαδή μπήκαν στο λαθρεμπόριο όπλων μέσω άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων και από εκεί πέρα συνδέθηκαν με προμηθευτές παρανόμων όπλων και απέκτησαν και γνώση για τις διαδρομές ε, και την υποδομή για να προχωρήσουν σε αυτό το έργο. Οι πολύ εγκληματικέ ομάδες που έχουν συνδεθεί ε, επίσης εμπλέκονται σε εκβιασμούς, λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ανθρωπίνων όντων, ε, διευκόλυνση παράνομης μετανάστευσης και ε, εξέπλημα βρώμικου χρήματος ε, και παραχάραξη χαρτονομισμάτων. Ειδικά όσοι κάνουν, ε, όσες ομάδες κάνουν βία εγκλήματα, όπως παραδείγματος χάρη ληστείες τραπεζών ή προβαίνουν σε βίες ενέργειες κατά άλλων αντιπάλων συμμοριών, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. και από ό,τι φαίνεται για αυτούς το λατρεμπόριο όπλων είναι κάτι το οποίο του δίνει την δυνατότητα να εγκληματίσουν. Οι συνεισφορέ από τα κράτη-μέλη μιλάνε για περιορισμένο ποσό που αφορά κυρίως ελαφρά όπλα. Η συλλογή των δεδομένων μας δεν έδειξε αύξηση στην, ε, ε, στο λαθρεμπόριο βαρέων όπλων. Βεβαίως ε, συχνά εκμεταλλεύονται αυτές οι ομάδες και τις αδυναμίες ε, στους ε, νόμιμες οδούς εμπορίας όπλων. Βλέπουμε ότι υπάρχει επίσης συσχετισμός ε, μεταξύ του λαθρεμπορίου όπλων και των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, γιατί και τα δύο αυτά ξεκίνησαν από τα Δυτικά Βαλκάνια και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Και επίση και η Τσεχία και η Σλοβακία έχουν αναφέρει ως χώρες πηγές για το λαθρεμπόριο όπλων. Οι βασικές πηγές παρανόμων όπλων ε, παραμένει επίσης οι, οι κλοπές διαρρήξεις, ε, νόμιμα όπλα τα οποία πολλούνται στην παράνομη αγορά και η, επαν, ε, η μετατροπή αχρηστευμένων πυροβόλων όπλων και αεροβόλων παρά το ότι, όπως είπα, είναι περιορισμένο το εμπόριο, βλέπουμε πως η διαθεσιμότητα των παρανόμων όπλων για τους βίους εγκληματίας είναι σοβαρή απειλή για το κοινό και τις διοκτικές αρχές. Μέχρι στιγμής η Europol δεν έχει ξεκινήσει κάποια επιχείρηση για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο όπλων απλούστατα γιατί δεν το έχουν ζητήσει οι διοκτικές αρχές των κρατών μελών. Ούτε έχει τεθεί ως προτεραιότητα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Europol ήδη έχει συσσωρεύσει γνώσεις και είναι έτοιμη να εμπλακεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη Ήδη επί σειρά ετών υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ, όπως η Task Force της Βαλτικής ε, και διάφορες άλλες ε, σχετικές δραστηριότητες για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Επίσης, ε, εξετάζοντας το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων, κοιτάμε και τις επιχειρήσεις που στηρίζουμε σε σχέση με το λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων. Ήδη έχουμε καθορίσει, ε, έχουμε βγάλει μια προειδοποίηση για την παράνομη χρήση από α, ε, συμμορίες πυροβόλων όπλων και προετοιμάζουμε άλλη μια προειδοποίηση. Επίσης, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την εσωτερική ασφάλεια προτείναμε στο Συμβούλιο για το 2014 να αποτελέσουν τα πυροβόλα όπλα έναν τομέα προτεραιότητας. Βεβαίω η Europol είναι έτοιμη για να σχεδιάσει μια ομάδα που θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα, όπως κάνουμε και με όλες τις άλλες προτεραιότητες που καθορίζει το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρίνη τώρα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ που καλέσατε την Επιτροπή να σας μιλήσει για την ε, κατάσταση που αντιμετωπίσουμε. Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν κοινό παρανομαστή στο οργανωμένο ε, έγκλημα. Αποτελούν άμεση απειλή στους Ευρωπαίους ε, πολίτες με ολέθρια αποτελέσματα όπως είδαμε στο, στην Ορβηγία ιδιαίτερα, στη Γαλλία ή εδώ και στο Βέλγιο. Πρόκειται για μία καθόλου καθησυχαστική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την Ιντερπολ, τα πυροβόλα όπλα χρησιμοποιούνται για... χρησιμοποιήθηκαν σε 245.000 δολοφονίες ανά τον κόσμο, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις πολιτικές ε, ή ένοπλες σειράξεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, διαπράχθηκαν πάνω από 5.000 δολοφονίες με πυροβόλα όπλα, δηλαδή το 20% όλων των ε, δολοφονιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της, του, των Ηνωμένων Εθνών της οργάνωσης UNODC. Γι' αυτό, όπως είχε πει ο πρώην Γενικός Γραμματέας ο Κόφι Ανάν το, στα Ηνωμένα Έθνη, ε, λειτουργούν σαν όπλα μαζικής καταστροφής. Γι' αυτό και έχουν προσελκύσει την προσοχή μας. Σε αντίθεση με τα ναρκωτικά ή τα παραχαραγμένα προϊόντα, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ' επανάληψη, όπως ε, είδαμε και στην περίπτωση των, ε, το, της περίπτωσης της Τουλούζης, όπου χρησιμοποιήθηκε ένα πυροβόλο όπλο που είχε κατασκευαστεί το 1944. Τι μας ενδιαφέρει λοιπόν. Μας ενδιαφέρει στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης το 2009 να τονίσουμε την χρήση των πυροβόλων όπλων που αποτελούν ε, μια πρόκληση ασφάλειας για, τα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των βαρέων πυροβόλων όπλων, ε, προσπαθώντας έτσι να καταπολεμήσουμε τη χρήση τους. Ε, πέρα από αυτή την πολιτική δέσμευση, πολλά έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία. Το Ηνωμένο ε, το... Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε, έχει εγκρίνει και έχει επικαιροποιήσει την νομοθεσία τη σε σχέση με την κατοχή, πώληση και μεταφορές όπλων μεταξύ κρατών μελών. Ε, το νομοθέτημα αυτό ενημερώθηκε το 2008, άρα μέχρι το 2014 θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν μία βάση δεδομένων σε σχέση με την κατοχή όπλων, νόμιμη κατοχή όπλων. Επίσης, η Επιτροπή έχει προτείνει ε, μία νέα νομοθετική ρύθμιση για το πρωτόκολλο κατοχής πυροβόλων όπλων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοιχνεύουμε την κατοχή των όπλων που εξάγονται και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε λοιπόν ώστε να συναφθεί, να συνταχθεί το πρωτόκολλο κατοχής πυροβόλων όπλων. Έχει επιτευχθεί πρόοδο σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή οι 18.000 αστυνομικοί, τελεωνιακοί και ελεγκτές συνόρων ε, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε 24ωρη βάση, ανοιχνεύοντας όπλα από το 2014. Επίσης, χρησιμοποιούμε την, ε, κοινή, το κοινό πλαίσιο ελέγχου στα σύνορα για να ανοιχνεύσουμε τη χρήση όπλων και τις αγωγές όπλων. Επίσης μιλάμε για τη, τους νέους οργανισμούς πραγματογνωμοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ε, ρόλο σε αυτό το φόρουμ βέλτιστων πρακτικών. Επίσης έχουμε επιταχύνει τη συνεργασία μας με τις χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Τα κράτη-μέλη και η Europol συνέχισαν να ανοιχνεύουν τους κινδύνους στα πλαίσια παράνομης εμπορίας όπλων από τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου, ε, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν 4 εκατομμύρια μη καταγεγραμμένα πυροβόλα όπλα και όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύραξης στα Δυτικά Βαλκάνια. Προσπαθούμε λοιπόν να προβούμε στη χαρτογράφηση αυτής της παράνομης δραστηριότητας και εμπορίας. Επίσης, η δήλωση των τυράννων τονίζει τη σημασία αύξησης ελέγχων και βελτίωσης της συλλογής στοιχείων και ανταλλαγής στοιχείων σε συνεργασία με την αστυνομία έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν αυτές οι χώρες με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως χρειάζεται περαιτέρω δραστηριότητα γνωρίζουμε ότι τα πυροβόλα όπλα δημιουργούν μεγαλύτερες βλάβες από ό,τι αρχικά νομίζαμε, γιατί χρησιμοποιούνται και από τους τομοκράτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Europol, οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν περισσότερα πυροβόλα όπλα παρά εκρηκτικά σε σχέση με το παρελθόν. Δυστυχώς αυτό γίνεται και στα εξωτερικά μας σύνορα από τις γείτονες χώρες όπου δεν υπάρχει στεναρός έλεγχος της αποθήκευσης αυτών των όπλων. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και δημιουργούν και διανέμουν όπλα χρησιμοποιώντας τα διάφορα εξαρτήματα τα οποία βρίσκουν από το διαδίκτυο και μπορούν να τα μετατρέψουν σε πολύ επικίνδυνα όπλα. Επίσης μπορούν να επανενεργοποιήσουν παροπλισμένα όπλα που βρίσκουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά στοιχεία είναι δυσέβρετα, αλλά γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των πυροβόλων όπλων στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπερβαίνει ο αριθμός αυτών, αυτός των καταγεγραμμένων όπλων που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί, όπως μας ε, ε, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο όπλων που χρησιμοποιούνται για τη θύρευση και το 2011 μόνο στη Γαλλία κατασχέθηκαν 3.910 πυροβόλα όπλα, δηλαδή 40% περισσότερο από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται για μια κερδοφόρα δραστηριότητα για τις εγκληματικές ομάδες που τις συνδυάζουν με την εμπορία ναρκωτικών. Η συνολική αξία του παράνομου εμπορίου σε πυροβόλα όπλα αποτιμάται σε 170, από 170 εκατομμύρια σε 320 ετησίως. Γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να συλλέξει στοιχεία για να μπορέσει να εξηχνιάσει το πρόβλημα. Πώς μπορούμε να κινηθούμε πέραν αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου που διοργάνωσε η DG Home το Νοέμβριο πέρσι, η Επίτροπος Μάλστρομ και ο Γενικός Διευθυντής Μανσερβίση αποφάσισαν να προβούν στη σύσταση μια task force. Έγιναν διάφορες πραγματογνωμοσύνες και ανταλλάχθηκαν απόψεις για τη χρήση των πυροβόλων όπλων. Μιλάμε για τεχνικές γλώσσες και πολιτική ε, κατανόηση του ζητήματος μέσα στα πλαίσια της ασφαλείας. Στόχος της Task Force είναι να ορίσει μια πολιτική που θα οδηγήσει σε ένα πακέτο χρήσης πυροβόλων όπλων μέχρι το 2015, ε, έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση αυτών. Γι' αυτό η Task Force ε, συντάσσει, ορίζει μία στρατηγική για να μειώσει τους κινδύνους από τη χρήση πυροβόλων για τους πολίτες και για να μειωθούν και τα κέρδη των εγκληματικών οργανώσεων. Η στρατηγική θα αποτελέσει αντικείμενο μιας ανακοίνωσης που θα εγκριθεί τον Οκτώβριο. Η ύψη τη σημασία είναι και η δημιουργία νέας νομοθεσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και ορισμός ενός συστήματος για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. Η πρόταση του Συμβουλίου μετά το πρωτόκολλο πυροβόλων όπλων των Ηνωμένων Εθνών είναι και το πρώτο που θα δημιουργήσει η Task Force. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να ελέγξουμε τη χρήση τους, να επιβληθεί ο νόμος και να μπορέσουν να δράσουν και οι ΜΚΟ. Μία βασική πτυχή των δραστηριοτήτων της ομάδας κρούσης είναι η πραγματική επικοινωνία με το κοινό για τους κινδύνους της χρήσης και παράνομης εμπορίας των πυροβόλων όπλων. Ε, επίσης γίνεται μία δημόσια διαβούλευση ε, μέσω του Your Voice in Europe. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη και τις οργανώσεις θυμάτων, μη κυβερνητικέ και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να απαντηθεί και το ερωτηματολόγιο ε, της Γενικής Διεύθυνσης Enterprise του 12 σε σχέση με τη χρήση πυροβόλων. Θα ενταχθούν όλα αυτά στην τελική ανακοίνωση της Επιτροπής. Το έγκλημα που σχετίζεται με τη χρήση πυροβόλων ε, έχει αυξηθεί και σχετίζεται με τη γενικότερη ατζέντα μας. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα επερχόμενα έτη. Επίσης ε, θα λάβουμε υπόψη και τις ε, προτεραιότητες αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν οι δημόσιες αρχές όλων των κρατών μελών να καταπολεμήσουν τη χρήση πυροβόλων αυτών. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Marini. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο κ. Γκολέτη. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Να σας μιλήσω για την επίσημη γαλλική αγορά την οποία γνωρίζω καλύτερα και όσα γνωρίζουμε για το λαθρεμπόριο όπλων. Για την επίσημη γαλλική αγορά μετά από διάφορες ρυθμίσεις υπό μεταρρύθμιση από το 1995 τόσο ευρωπαϊκές όσο και γαλλικές η αγορά έχει επαγγελματικοποιηθεί και μοιράζεται σε διάφορα σημεία πώληση πολύ πιο ελεγμένα. Στη Γαλλία ο, των διαδικασιών για να έχει κανείς ένα ε, κατάστημα όπλων ε, μείωσε, οδήγησε στη μείωση των ε, καταστημάτων αυτών. Έχουμε λιγότερο από χίλια καταστήματα σήμερα. Χρειάζονται τέσσερι άδειε για να έχει κανείς το επάγγελμα, να ασκεί το επάγγελμα του οπλουργού. Μια έγκριση που σχετίζεται με το κατάστημα ε, το ίδιο της πώληση, μια έγκριση για τις, ε, τα όπλα κατηγορίας C και D και για, άλλη άδεια για τα όπλα κατηγορίας Α και Β που ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια. Τέλος, έγκριση για τον υπεύθυνο του καταστήματος, ένα είδος διπλώματος πτυχίου ε, οπλουργού που ανανεώνεται επίσης κάθε 10 χρόνια. Έτσι έχουμε τελείως ε, απομακρύνει τους απαταιώνες από αυτό το επάγγελμα. Θα πρέπει να προσθέσουμε και απόλυτα διασυνδεδεμένους φακέλους για όλους τους εμπλεκόμενους. Έχουμε στη Γαλλία ένα φάκελο για την έγκριση της αδείας κυνηγίου που συγκρίνεται με τις απαγορεύσεις κατοχής όπλου. Ας πούμε, αν ένας άνθρωπος ε, απαγορεύεται να έχει την κατοχή του όπλου αμέσως το βλέπουμε. Επίσης, συνδέεται με το, φυσχέ, με το ε, αρχείο ε, απαγόρευσης κατοχής όπλου. Ε, υπάρχει και σύνδεση ανάμεσα στις διάφορες διοικήσεις ε, της αστυνομίας, ε, της, της δικαιοσύνης, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουν περάσει από ψυχιατρία ή είχαν προηγούμενα ψυχιατρικά προβλήματα. Και τέλος έχουμε για όλα τα όπλα κατηγορίας α, β, γ και δ, μητρώα για το, αυτά που κυκλοφορούν ή ε, πολλούνται στη Γαλλία μέσω αυτού του συστήματος αρχείων. Αυτό το σύστημα λοιπόν αρχείων καθιστά στο εσωτερικό της Γαλλίας για την επίσημη αγορά την ε, κυκλοφορία ενός όπλου γιατί ε, παρακολουθείται από το α μέχρι το ω. Ένας νέος δόμος ψηφίστηκε Δε το 2012 σχεδόν ε, ομόφωνα από το ε, Εθνοσυνέλευση είναι σπάνιο αυτό να υπερψηφιστεί από τη δεξιά και την αριστερά ομόφωνα σχεδόν ένας νόμος ο οποίος επιβαρύνει πάρα πολύ την ποινική πτυχή της ε, κατοχής και παράνομης χρήσης ή εμπορίας όπλου για όλες τις κατηγορίες. Το εμπόριο όπλων ακόμα και για τις πιο απλές κατηγορίες δεν είναι απλό παράβαση αλλά είναι ε, παράπτωμα ε, σοβαρό. Και για όλες τις κατηγορίες ε, θα υπάρξουν διατάγματα τα οποία θα εκδοθούν πριν από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Η μεταγραφή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα ολοκληρωθεί πριν η Γαλλία είχε οκτώ κατηγορίες, ενώ τώρα θα έχουμε τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή ε, Οδηγία Α, Β, Γ και Δ, όπου γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στα στρατιωτικής χρήση όπλα και τα πολιτικής χρήση όπλα το κείμενο αυτό θα απλοποιήσει βασικά τη ζωή 1,5 εκατομμυρίων νομίμων χρηστών όπλων στη Γαλλία και την ζωή του διοικητικού μηχανισμού που μέσα σε μια περίπλοκη σχετικά νομοθεσία δυσκολευόταν να εντοπίσει κάθε φορά τα όπλα τα όπλα κατηγορίας Α, ε, Β στη Γαλλία μπορούν να αγοραστούν μόνο από σκοπευτές μετά από άδεια. Οι άδειες ε, για λόγους αμήνης είναι πολύ σπάνιες και χωρούνται μόνο υπό συγκεκριμένη άδεια και χρειάζεται περίπου τέσσερις μήνες για να πετύχει, πάρει κανείς άδεια κατοχής όπλου. Πολύ λίγες άδειες ε, χορηγούνται για λόγους αμυντικούς στη Γαλλία για τα όπλα σε κατηγορία C και D, ε, αυτά μπορούν να τα έχουν μόνο κυνηγοί μετά από ε, συγκεκριμένες εξετάσεις που τους γίνονται με ε, ιατρικές εξετάσεις και για τους σκοπευτές χρειάζεται άδεια σκοποβολής με συγκεκριμένες ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο ανανεώνεται ετησίως. Ε, και για όλα τα όπλα κατηγορίας Β, αυτά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε συγκεκριμένες θηρίδες ή να είναι ε, δεμένα με αλυσίδα και τα πυρομαχικά τους θα πρέπει να φυλάσσονται ξεχωριστά. Κανένα φωνικό όπλο δεν μπορεί να πολιθεί δε στη Γαλλία σε ανθρώπους που δεν είναι κυνηγοί ή σκοπευτές. <coughs> Απαγορεύεται δε η πώληση σε ανήλικους. Αυτά λοιπόν για την επίσημη αγορά. Τώρα, για το λαθρεμπόριο όπλων, όπως για το, για το λαθρεμπόριο, είναι αδύνατο να έχουμε στοιχεία και ακριβή επειδή είμαστε υπεύθυνοι για την επίσημη αγορά, ίσω να μην είμαστε πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε για την παράνομη αγορά. ίσως οι ε, ε, ε, τήρησης της τάξης να είναι σε καταλληλότερη θέση, αλλά συμμετέχουμε σε συνεδριάσεις όπου κάνουμε ανταλλαγέ σε πληροφοριών. Πρόσφατες πληροφορίες από τη Γαλλική Αστυνομία, οι κατασχέσεις όπλων είναι σταθερές και μικρές εδώ και πολλά χρόνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 3.910 όπλα κατασχέθηκαν το 2010 Συγγνώμη, το 11 ε, διορθώνει ο μιλητής, σε σχέση με το 2010 έχουμε αύξηση 44%, αλλά είναι πολύ σχετικά τα πράγματα γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ περίπλοκη. Έχουμε επανέλθει στο νούμερο του 2004 που είχαμε 4.400 ε, κατασχέσεις και το 2008 4.000. Το μερίδιο των Καλάσνικοφ ανάμεσα σε όλα αυτά τα όπλα είναι πολύ μικρό. Νέο γεγονός είναι ότι οι τρομοκράτες ή οι υλοποδίτες χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά ε, όπλα πολέμου τύπου Καλάσνικοφ που απαγορεύονται από την ε, οδηγία του 93 στην Ευρώπη. 164 τέτοια μοντέλα ε, κατασχέθηκαν το 2011 ενώ ήταν 80 το 10 και 67 το 9. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δούμε από πού προέρχονται αυτά τα όπλα αλλά κυρίως προέρχονται από τα Βαλκάνια. Ένα μεγάλο κομμάτι των όπλων που κατάσχονται στη Γαλλία είναι όπλα από την τελευταία πόλεμο κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν ε, ε, μάχες στα εδάφη αυτά, όπου πολλές φορές ε, ρίχτηκαν με αλεξίπτωτο τα όπλα εκεί και ε, εγκαταλείφθηκαν εκεί από τα υπόλοιπα μέρη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια καταστολής του λαθρεμπορίου όπλων που να ενταχθεί βέβαια στη... και να ενταχθεί στην πάταξη του λαθρεμπορίου όπλων, ναρκωτικών ε, και έργων τέχνης. Το 2009 ε, διαπιστώσαμε την ε, κυκλοφορία όπλων πολύ πιο εξελιγμένων, αλλά η κατάσταση δεν είναι δραματική όσον αφορά το λαθρεμπόριο. Κατά τη γνώμη του Αρμοδίου ε, υπήρξε μια άφηξη όπλων, πολεμικών όπλων, μετά από το τέλος του πολέμου το 2000, το 1991 και όμως η πηγή αυτή έχει πια ε, στερέψει. Οι στατιστικές για τα όπλα πολέμου δεν αναφέρουν λεπτομέρειες, αλλά η αύξηση της χρήσης αυτής ε, θεωρείται μικρή ε, από τον Υπουργό Εσωτερικών, το οποίο οι υπηρεσίες τίμησαν το 2012 ότι παρά την μεγάλη διάδοση της χρήσης του Καλάζνιχοφ. Αυτό το όπλο είναι δύσκολο να το αποκτήσει κανείς, δεν είναι πολύ εξαπλωμένη χρήση του και κυρίως χρησιμοποιείται από τους ε, ε, μεγάλους, ε, από μεγάλες οργανωμένες ομάδες. Το Το 2011 ε, ε, είχαμε 1.200 ανθρωποκτονίες και το 2012 1914. Γενικά έχουν μειωθεί ανθρωποκτονίες και γενικά τα όπλα είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για το 20% των ανθρωποκτονιών. Οι ανθρωποκτονίες κατά τη διάρκεια ληστείων μειώνονται βασικός ε, αίτιο είναι η, ε, τα ε, εγκλήματα πάθους είτε η, το οργανωμένο έγκλημα. Έχουν χρησιμοποιηθεί δε όπλα κατά τη διάρκεια διαφόρων ε, μαχών ανάμεσα σε ομάδες ε, εγκληματιών. Στην ε, δολοφονίες του λουζης χρησιμοποιηθηκαν χρησιμοποιήθηκαν ένα S10, ένα ούζι, το S10 και το ούζι απαγορεύονται από, τελείως από, εντελώς από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δεν ήταν καταγεγραμμένα δε αυτά τα όπλα, δεν είχαν κλαπεί από την επίσημη αγορά, ούτε είχαν εξαφανιστεί από αυτήν. Άρα λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το λαθρεμπόριο όπλων βασικά γίνεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος στα σύνορα και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχουν τόσες σχέσεις ανάμεσα στην επίσημη αγορά όπλων ε, και το λαθρεμπόριο όπλων όσο υπάρχει σχέση ανάμεσα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ε, τα ε, επίσημα φαρμακεία. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκολέτη. Κύριε Γιακολίνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ακούσαμε και τις τρεις παρεμβάσεις των εισηγητών. και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και το πάνελ ε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει ε, γνωρίζω τα αυτά αποτελέσματα τα οποία μας παρουσίασε, παρουσίασε και ο κύριος ε, Μαρίνη. Το θέμα της παρά, το παράνομου εμπορίου των όπλων είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, αφορά και τρομοκρατικές οργανώσεις και το, από τον Ιανουάριο υπάρχει αυτή η task force έτσι ώστε να υπάρχει και ολοένα και μεγαλύτερος έλεγχος. Έχει μεγάλη σημασία η ανιχνευσιμότητα εμείς προβλέπουμε ένα τσιπάκι για τα όπλα και ασχοληθήκαμε και με το παράνομο εμπόριο των όπλων. Και οι τρεις παρεμβάσεις και οι τρεις εισηγήσεις ε, αφορούν μία καλύτερη οριοθέτηση του θέματος, ιδιαίτερα ως προς τις άδειε που χορηγούνται. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανακράτος και είπαμε σήμερα το πρωί ότι θα πρέπει να μειωθεί και ο γραφειοκρατικός φόρτος. Και μέσα στα πλαίσια της εμπορίας Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα σωστότερο πλαίσιο αδειοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζεται και από την Europol όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την ανακύκλωση βρώμικου χρήματος. Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές στον εκπρόσωπο της Europol θα ήθελα να υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Είπατε ότι μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν απαντήσει ή θεώρησαν ότι ε, δέχονται κάποια απειλή. Ποια είναι αυτά τα τρία κράτη που δέχονται απειλές. Πρόκειται για πρώην ανατολικά κράτη φαντάζομαι. Εμείς στην Κορσική και στη Μασαλία αντιμετωπίζουμε μεγάλους ε, κινδύνους. Υπάρχουν νεκροί και πολλές φορές χρησιμοποιούνται όπλα σνικόφ. Δεν υπάρχει μεγάλο εμπόριο των Καλάσνικοφ. Είναι περιορισμένο. προέρχεται από πρώην εμπόλεμες ε, περιοχές, αλλά νομίζω ότι μπορεί να περιοριστεί. Είπατε ότι ως προς τα ελαφρά όπλα δεν υπάρχει ε, μεγάλο εμπόριο. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Μας είπατε επίσης ε, ότι υπάρχει ε, νέα χρήση όπλων που ε, θεωρούνται παροπλισμένα. Το 2008 στην οδηγία για τα όπλα ασχοληθήκαμε με αυτά τα όπλα που είχαν υποτίθεται εξουδετερωθεί. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με την οδηγία του 8. Μας είπατε ότι υπάρχουν, ε, υπάρχει και χρήση ορισμένων... Ε, ορισμένων αεροβόλων. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν αυτά τα και να αγοραστούν παράνομα αυτά τα αεροβόλα. Μπορείτε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες. Κύριε Μαρίνη, είπατε για τέσσερα εκατομμύρια όπλα που έχουν καταγραφεί. Τέσσερα εκατομμύρια, καλά άκουσα. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Μαρίν. Dans toute l'Union Européenne. Α, μόνο στη Γαλλία. Μόνο στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τα τέσσερα εκατομμύρια. Μόνο στη Γαλλία. γιατί υπάρχουν 7 εκατομμύρια κυνηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλώ για αθλητικές δραστηριότητες, σκοποβολή και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε για 7 εκατομμύρια ε, κυνηγούς ε, που συμμετέχουν σε κυνήγι διάφορες εποχές, όταν κυνηγάνε αγριογούρουνα ή σε άλλες, άλλες εποχές, καταλαβαίνετε ότι έχουμε να κάνουμε 14 εκατομμύρια όπλα. Μπάς περιπτώσει δεν είναι δολοφόνοι. Δεν σας μιλώ για, το, για τις αθλητικές δραστηριότητες, για τη σκοποβολή, για τα Ολυμπιακά αθλήματα. Πρόκειται για θέμα ασφάλειας. Όταν ε, εγώ μεταβαίνω στην Ισπανία, στη Φιλανδία, ε, για κυνηγετικούς σκοπούς, φεύγω από τις Βρυξέλλες, μεταβαίνω στη Μαδρίτη και το όπλο ελέγχεται και από τις Βρυξέλλες και από τη Μαδρίτη και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αυτό αφορά και τους κυνηγούς και τους αθλητές που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας. Θα πρέπει να σταματήσει το εμπόριο των ε, Καλάσνικοφ, των αεροβόλων. Δεν μιλάμε εδώ για τους κυνηγού. ή για εκείνους που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο εισηγητής μίλησε για βελτιωμένη ανιχνευσιμότητα. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αναχαιτήσει την ελεύθερη κυκλοφορία υλικού. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Thank you very much. Yes. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Όταν ανέφερα τις τρεις χώρες αυτές. Ε, στόχος ήταν να τα θέσω αυτά σε ένα πλαίσιο των απειλών που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορώ να σου πω ποιες είναι οι χώρες, αλλά αναφέρονται στην έκθεσή μας. Αλλά Λίγε χώρε το έχουν ω υψηλή απειλή. Τώρα για το ερώτημα για τα Καλάσνικοφ και τη μετατροπή όπλων και αεροβόλων. Έχουμε και παραδείγματα περιπτώσεων που έχουμε δει στη δουλειά μας. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Μαρίνη, δεν έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό η Europol θα ξεκινήσει μια λεπτομερή ανάλυση κινδύνου. Βεβαίω το οργανωμένο και σοβαρό έγκλημα αφορά πολλά τέτοια φαινόμενα και δεν μπορούμε με λεπτομέρεια να καταγράψουμε κάθε έγκλημα που διαπράττουν οι συμμορίες. Οπότε, όπως είπα, θα μας απασχολήσει στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου μια αξιολόγηση κινδύνου για το λαθρεμπόριο όπλων και θα ξέρουμε άρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ε, θα το δούμε τώρα λεπτομερώς και μετά μάλλον θα μπορέσουμε να σας δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει σε αυτή την ε, εγκληματική αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Θα ήθελα να σας καθησυχάσω όλους ε, η Επιτροπή δεν θέλει να θίξει τους νόμιμους κατόχους ε, πυροβόλων όπλων, αθλητικές οργανώσεις, αθλητές, κυνηγού κλπ. Θα ήθελα να σας πω πώς ε, θέλουμε να δράσουμε και να οργανώσουμε τη δραστηριότητά μας. Εάν δούμε ότι, για παράδειγμα, γίνονται πολλά ε, ατυχήματα στους δρόμους ενός άξονα, δεν σημαίνει ότι σταματά η δραστηριότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά αντιμετωπίζονται in situ τα ατυχήματα, οι οδικές αρτηρίες δηλαδή. Δεν ε, θα πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό κάθε φορά, αλλά να καλύψουμε τα νομικά κένα που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, δεν γνωρίζα εγώ τη νέα ε, γαλλική νομοθεσία και με εκπλήσει το πώς αντέδρασε η Γαλλία, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με την ιατρική γνωμάτευση και πιστοποίηση, δεν προαπαιτείται από όλε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μορφή διασφάλισης έτσι ώστε αυτός που, ζητήσει, που ζητά την άδεια να ξέρουμε ότι γνωρίζει τι κάνει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα αεροβόλα. Μίλησα σε ένα γερμανό κατασκευαστή, με ένα γερμανό κατασκευαστή, ο οποίος μου είπε ότι ότι ό,τι προέρχεται από την Τουρκία παρουσιάζει προβλήματα κατασκευαστικά ελαττώματα δηλαδή. Εάν ε, προσπαθήσουμε λοιπόν να μετατρέψουμε ένα όπλο σε πυροβόλο, τότε κινδυνεύει να εκραγεί. Ότι προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, ενέχει κινδύνους. Υπάρχουν πολλά νομικά κενά τα οποία θα πρέπει να καλύψουμε. Γι' αυτό και μιλάμε για τους ε, διάφορους ε, φορείς, ερευνητές, ε, πολίτες κλπ. Έτσι ώστε να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να είναι αποδεκτές για όλους. Για να αυξήσουμε την ασφάλεια χωρίς να επιβαρύνουμε όμως την νομοθεσία και να επιβάλλουμε πράγματα που δεν είναι κατανοητά. Να πάρουμε όμως ό,τι είναι καλύτερο σε κάθε κράτος. Αυτό, είναι το μέλημά μας. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα στα, στη Γαλλία σε σχέση με την εξουδετέρωση όπλων. Υπάρχει μια επίσημη, ένας επίσημος φορέας, δεν μπορεί να το κάνει ένας οπλουργός. Και αυτό είναι κάτι πολύ καλό γιατί υπάρχει ένας ε, ελεγκτικός μηχανισμός αυτής της εξουδετέρωσης. Το ίδιο αφορά και όπως είπε και ο κύριος Μαριάννη και για τα όπλα γενικότερα. des cargaisons entières. Dans Αυτά τα όπλα τύπου alarm, τα οποία κατασκευάζονται εντός και εκτός Ευρώπης, ε, είχαμε μία τέτοια κατασκευή, τέτοιες κατασκευές ε, στην Τουρκία, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι μικροεγκληματίες. Και τα όπλα τύπου αλλά επίσης θα πρέπει να δοκιμαστούν έτσι ώστε να μην διατρέχει κανείς κανένα κίνδυνο. Άρα είμαστε σίγουροι για το τι βάζουμε στην αγορά, τι κυκλοφορεί στην αγορά. Eh Νομίζω ότι μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην κυρία Αλφάνο η οποία επέστρεψε από μια άλλη συνεδρίαση όπου βρισκόταν. Allora, riprendiamo i lavori. Io Ζητώ συγγνώμη για την απουσία μου και ευχαριστώ τη Βερονίκ που ανέλαβε την Προεδρία. Είχαμε και τις ε, ε, ε, εργασίες, είχα και ήμουν σκιώδη σε μία άλλη επιτροπή και έκθεση. Τώρα περνάμε στο δεύτερο κλάστερ E Σε σχέση με τον έλεγχο στα σύνορα, θα ακούσουμε τον Κλάους Ρέσλερ από τη Frontex που θα μας μιλήσει για τον, για τον ε, συντονισμό στα σύνορα από πλευράς της Frontex. Τον ε, κύριο Παϊγκοζίνας που θα μας μιλήσει για τον ε, έλεγχο στα λιθουανικά σύνορα, τον κύριο Μπαρτονομία Ιτσίκ, ο οποίος είναι υπεύθυνος ε, διευθυντής του Business Development Northeast Europe και θα μας μιλήσει για τον ε, έλεγχο στα σύνορα, ιδιαίτερα της Πολωνίας και τον Τέχρο Ραγιάλα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος από τις φιλανδικές αρχές. Ο κάθε εισηγητής έχει 15 λεπτά. Ο κύριος Κλάους Ρέσλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ που καλέσατε την Frontex για να συνεισφέρουμε στο θέμα αυτό. Η αποστολή της Frontex είναι ε, ο αποτελεσματικό έλεγχος των συνόρων και η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Γι' αυτό ο στόχος των κοινών επιχειρήσεων που θα γίνουν στα ανατολικά σύνορα το 2013 είναι να αυξηθεί η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στα χερσαία σύνορα και το σχετικό οργανωμένο έγκλημα, να ενισχυθεί η συνεργασία των υπηρεσιών και με τις γειτονικές τρίτες χώρες. Να αναπτύξουμε κοινέ ομάδες και να έχουμε κάποιες επιχειρήσεις σε σχέση με την ένταξη της Κροατίας και να δούμε τι θα γίνει με την ένταξη της, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ζώνη Σέγγεν. Το 2010 είχαμε την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου και έχουμε τρεις εξελίξεις σε σχέση με αυτό. Πρώτα απ' όλα, η διασυνοριακή ροή επιβατών συνεχίζει να αυξάνεται το 2012, κυρίως στα πολωνορωσικά σύνορα, στα νορβηγορωσικά ε, σύνορα και στα σύνορα με την Πολωνία και ε, πολωνιας Και βέβαια αυτό οφείλεται και στις οικονομικές εξελίξεις ε, στη Ρωσική Ομοσπονδία και πρέπει να σκεφτούμε πως μιλάμε για χερσαία σύνορα 6.000 χιλιόμετρων, αλλά ε, είναι μόνο 2% των ε, παρανόμων διελεύσεων των σύνορων, αλλά 35% των απαγόρευσης, των απαγόρευσεων εισόδου. Η αύξηση των επιβατικών ροών οφείλεται σε περισσότερες διελεύσεις για λόγους εμπορίου και σε περισσότερες θεωρίες των Αυτό σημαίνει περισσότερες ευθύνες των συνοριακών φυλακίων και αυξάνεται ο κίνδυνος κατάχρησης ε, των νομίμων οδών ε, διελεύσεως ε, αντί για να αυξάνεται ο αριθμός των παρανόμων διελεύσεων. Μια δεύτερη εξέλιξη είναι το λαθρεμπόριο αγαθών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε δείχνουν πως το λαθρεμπόριο αγαθών είναι μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των συνόρων. Μιλάμε δηλαδή για προϊόντα καπνού, βενζίνης και χάνονται έτσι πάρα πολύ ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Επιπλέον, οι διασυνοριακές εγκληματικέ δραστηριότητες ε, φορούν την δυνατότητα να περάσουν κλεμμένα οχήματα και πιθανώ και ναρκωτικά. Το λαθρεμπόριο δεν αφορά μόνο βεβαίω τα φυλάκια τα συνοριακά, αλλά όλα τα χερσαία σύνορα. Και η τρίτη μεγάλη εξέλιξη είναι η αύξηση των ροών παράνομης μετανάστευσης που καταγράφηκε το 2012 και φαίνεται στις παράνομες διελεύσεις από τα χερσαία σύνορα και από τις αρνήσεις διέλευσης ε, και από τις ανιχνεύσεις ε, κατά την έξοδο. Η ανάλυση κινδύνου της ε, Frontex και η σχετική ετήσια έκθεση που έγινε σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη στο δίκτυο ανατολικών συνόρων βλέπει τέσσερις κινδύνους. Ο πρώτος είναι ο κίνδυνος λαθρεμπορίου, προϊόντων καπνού, προϊόντων βενζίνης, ναρκωτικών και αυτοκινήτων. Το δεύτερο αφορά την παράνομη μετανάστευση από χώρες μη ε, της, ε, από χώρες μη πρώην Σοβιετικής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της ε, απάτης σε σχέση με τα έγγραφα, πλαστογράφηση ε, βίζας ε, και λοιπές απάτες με έγγραφα. Το άλλο είναι η παράνομη μετανάστευση από τις χώρες της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών της Γεωργίας συμπεριλαμβανομένης και εδώ πέρα έχουμε βεβαίως παράνομη χρήση εγγράφων και ο τέταρτος κίνδυνος που σχετίζεται με αυτό είναι η κατάχρηση που γίνεται στους, ε, στις νόμιμες οδούς ε, διέλευσης, δηλαδή άνθρωποι που ζητάνε άσυλο ή άνθρωποι που μπαίνουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, ξεπερνάνε την διάρκεια παραμονής τους και με τους ανοιχνεύουμε συχνά όταν βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υψηλό αριθμός ανείχνευση οφείλεται επίσης και στους αποτελεσματικού ελέγχους και στην παρουσία ειδικών και στι αυξήσει ε, των δυνατοτήτων των αρχών ελέγχου των συνόρων στα ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι κοινέ επιχειρήσεις της Frontex του 2012 και 2013 στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της ε, παράνομης ε, μετανάστευσης με ε, πολλές στοχευμένες επιχειρήσεις. Η πρώτη και μεγαλύτερη είναι τα σημεία επαφής που, όπου επιλέγουμε βεβαίως να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία των συνόρων. Και αυτό σημαίνει βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε τις πλατφόρμες συντονισμού για να προχωρήσουμε σε στοχευμένες δραστηριότητες, κυρίως μέσω της ανάπτυξης ειδικών στον έλεγχο των συνόρων, των εγγράφων και από άλλα κρατημέλη, για να ενισχυθεί έτσι η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και χωρών Σέγγεν, για να υπάρξει επαγγελματική βοήθεια, να ανταλλάσσουμε ε, όπως είπα, εμπειρίες ε, και να προσπαθήσουμε να επιτηρήσουμε τα σύνορα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των σύνορων. Όσον αφορά την εφαρμογή, κάποια σημεία είναι μονίμως σημεία εστιασμού, κάποια άλλα προσωρινά. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν. Το 2012 προσθέσαμε κάποια από αυτά. Έχουμε 23 κράτη-μέλη που συμμετέχουν από αυτά, 12 ε, φιλοξενούν τα σημεία αυτά ε, που εστιάζουμε. Έχουμε αναπτύξει πάνω από 350 ειδικού ε, μονάδες θερμικής όρασης, σκύλους και φορητά εργαστήρια. Επίσης, ε, λόγω του προβλήματος Ελλάδας έχουν επηρεαστεί οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ειδικά τα χερσαία σύνορα Ουγγαρίας, Σερβίας ε, και Αλβανίας. Θα συνεχιστούν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις και στα ανατολικά χερσαία σύνορα το 2013 και πάλι όπως σας είπα 12 κράτη-μέλη και χώρες Σέγγεν από την Νορβηγία στο βορρά ε, ε, αναπτύσσουν ε, τέτοιες δυνάμεις και επιχειρήσεις έλεγχου των συνόρων και η δεύτερη, η δεύτερη κοινή επιχείρηση είναι η επιχείρηση συντονισμού. Σημαίνει πως κάποια τέτοια σημεία υπάρχουν μεταξύ δύο χωρών μη κρατών μελών, π.χ. στα σύνορα Κροατίας και Σερβίας, μέχρι να ενταχθεί η Κροατία βεβαίως, ή στα σύνορα Σερβίας και ε, της ε, Πούγουδουμού. Και ο επιχειρησιακός στόχος είναι να έχουμε ένα σύστημα άγγελης προειδοποίησης για να έχουμε επιχειρησιακές πληροφορίες για τις μελλοντικέ τάσεις παράνομης μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Όπως είπα, δεδομένη της ένταξης της Κροατίας, στηρίζουμε αυτή τη στιγμή την Κροατία για να ευθυγραμμιστούν πρακτικές των κρατών μελών για να καταλήξουμε σε κοινέ επιχειρήσεις. Το 2012 το έργο αυτό ε, διεξήχθη για 8 εβδομάδες και το 2013 προβλέπεται να ε, να διεξαχθεί πέντε φορές σε διαφορετικά ε, σημεία των σύνορων θα έχουμε σχεδόν 45 εβδομάδες εφαρμογής. Στα εξωτερικά χερσαία σύνορα θα εφαρμόσουμε ξανά την κοινή επιχείρηση Δίας για να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος παράνομης μετανάστευσης στα χερσαία σύνορα, να ενισχυθεί η συνεργασία των υπηρεσιών και με τις χώρες εκτός Ένωσης μέσω της ανάπτυξης των κοινών ομάδων ελέγχου συνόρων και εναρμόνισης της ανάπτυξής τους με τα σημεία εστιασμού. Το 2013 θα έχουμε μια φάση τεσσάρων εβδομάδων για τα χερσαία σύνορα και επιπλέον σε σχέση με την ενίσχυση των αεροπορικών σύνορων θα εφαρμόσουμε το πιλωτικό σχέδιο Ρήγα για να αυξηθούν οι γνώσεις των συνοριοφυλάκων για τις δραστηριότητε των διαφόρων δικτύων στα αεροδρόμια, να ενισχυθεί η υπηρεσιακή συνεργασία και να υπάρξει βεβαίω και καλύτερη εκπαίδευση για τη συλλογή πρώτων αποδεικτικών στοιχείων στα σύνορα. Το 2013 θα εστιάσουμε ειδικά στα παιδιά με στόχο να βρούμε τα κενά στις διαδικασίες ε, για τα παιδιά που χρειάζονται προστασία στα εξωτερικά αεροπορικά σύνορα, να συλλέξουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, και να υπάρξει ευαισθητοποίηση για τα παιδιά που ρίζουν προστασία. Με αυτές τις στοχευμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες, πέρα από την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση του δικτύου για τα ανατολικά σύνορα, θεωρούμε πως θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια αντίληψη της κατάστασης στα ανατολικά μας σύνορα και να στηρίξουμε τις αρχές των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο και να μειώσουν τους κινδύνους που ανέφερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα δίνουμε το λόγο στην κυρία Βιζάντα Βαζίνες Βίτσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για που μου δίνετε το λόγο και που με καλέσατε να μιλήσω σε αυτή την Επιτροπή. Θα μιλήσω σύντομα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα ανατολικά σύνορα και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Θα σας μιλήσω σύντομα λοιπόν για το εύρος του προβλήματος, για την απάντηση, την ανταπόκριση και τις πιθανές λύσεις. υπάρχουν ε, ε, παρεπιπτώσεις από την ε, επίσημο αγώνα κατά του λαθρεμπορίου ζυγάρων. Θα σας απαντήσω σε λίγο. Βασικά, λοιπόν, τα τσιγάρα περνάνε από τη Λιθουανία, από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξανόμενη απειλή προέρχεται από την πλευρά της Λευκορωσίας, όπου υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ε, ε, τσιγάρων που παράγονται στη Λευκορωσία από το 2010, κάπως ε, μειώθηκαν γιατί υπάρχουν και τσιγάρα που κατασκευάζονται στη θύλακα του Καλίνικραντ. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα ελεύθερου τσιγάρων από την Ρωσία μέσω της Λετωνίας ή της Λιθουανίας και των ε, συνόρων με τη Λευκορωσία. Ε, μπορείτε να δείτε έναν από τους κύριους επιταχυντές ε, του λαθρεμπορίου είναι η διαφορά της τιμής και το πιθανό κέρδος που μπορεί να έχει κανείς από την διάπραξη αυτού του κλίματος. Μέχρι και 1000% κέρδος μπορεί να έχει κανείς. Η πρόσφατη οικονομική κρίση καθώς και το υψηλό επίπεδο ανεργίας συμβάλλουν στην αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Τα κέρδη δε αυτών των οργανωμένων ε, ομάδων εγκλήματος είναι ε, το, βασικό βασική έλξη που ασκεί το λαθρεμπόριο αυτό. Εδώ βλέπετε ότι υπήρξε σημαντική μείωση στις κατασχέσεις τσιγάρων λόγω του ότι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο μεγάλες εγκληματικέ οργανώσεις αλλά και διάφορα φορτία του καπνού που προορίζονταν προς το παράνομα εργοστάσια που κατασχέθηκαν στην Πολωνία. 70 τόνοι ακατέργαστου καπνού κατασχέθηκαν ως αποτέλεσμα κοινών ερευνών του ε, αστυνομίας της Πολωνίας καθώς και των ε, γερμανικών ε, τελωνίων των μονάδων δίωξης εγκλήματος αυτών θα σας περιγράψω τη διαδικασία μιας από αυτές τις ε, εγκληματικές ε, ομάδες. Η ομάδα δίωξης εγκλήματος ε, των τελωνίων της Λιθουανίας δίωξε μια εγκληματική ομάδα. Όπως βλέπετε κατασχέθηκαν εκατομμύρια τσιγάρα και πολλά άτομα ε, διώχθηκαν στη Λιθουανία, Πολωνία και ε, Γερμανία. 50 άνθρωποι. Τώρα, το 2010, μετά από αίτημα των ε, τελωνίων της Λουθανίας και της μονάδας δίωξης εγκλήματος, ξεκίνησε μια ε, συντονιστική συνεδρίαση της Όλαφ, οι αρμόδιες αρχές ε, της Πολωνίας, της Γερμανίας επίσης συμμετείχαν και ξεκίνησαν σχετικές έρευνες που οδήγησαν στα αυτά τα αποτελέσματα στις κατασχέσεις και στις συλλήψεις στην Πολωνία, τη Γερμανία και τη Λιθουανία. Εδώ έχετε κάποιες εικόνες από τις κατασχέσεις. Όπως βλέπετε έχουμε, ε, τα, υπήρχαν παράνομα αγαθά τα οποία ε, περνούσαν ως εμπορεύματα. Στις 6 Απριλίου του 2011, επί τη βάση πληροφοριών που συλλέχθηκαν ε, μέσω των έρευνών, Με τη βοήθεια της ειδική ομάδας κατά της τρομοκρατίας της αστυνομίας της Λιθουανίας, καθώς και της ειδική μονάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, συνελήφθησαν οι πρώτοι ύποπτοι, καθώς και ε, υπάλληλοι που ήταν ύποπτοι για συνεργασία και διαφθορά. Αυτή η υπόθεση μάλιστα δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Θα περάσει από το δικαστήριο, θα εκδικαστεί τον Ιούνιο φέτος, 18 υποθέσεις που αφορούν λαθρεμπόριο τσιγάρων έχουν εκδικαστεί από το 2009 όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη έρευνα. Ε, όταν ε, ο αγώνας, ε, η, μάχη γίνεται πιο αποτελεσματική, κατάσχονται περισσότερα τσιγάρα, τσιγάρα και εν γέννη ε, αυξάνονται οι δαπάνε σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τα κατασχεμένα τσιγάρα σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφούν και άρα σημαίνει και περισσότερες δαπάνες για τα τελωνία. Έχουμε συγκεκριμένες αποθήκες που είναι υπεύθυνε, ε, έχουμε συγκεκριμένα μάλλον ε, μονάδες των τελωνίων που είναι υπεύθυνε για τη μεταφορά, την αποθήκευση και την καταστροφή των ε, τσιγάρων. Και εδώ έχουμε μόνο ένα παράδειγμα, περίπου 700.000 ευρώ είναι η ετήσια δαπάνη των λιθουανικών τελωνίων για τη διατήρηση αυτού του είδους των αποθηκών τύπου F, μόνο για τσιγάρα δηλαδή. Λίγα λόγια για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή την εικόνα, πέρυσι έχουμε μία κινητή μονάδα ακτινών Χ και μία σταθερή. Και φέτος έχουμε τρεις κινητές μονάδες. Μία στα σύνορα με τη Λευκορωσία, τη βλέπετε δεξιά, και μία στα σύνορα με την περιοχή του Καλίνιγκραντ που ανήκει στην ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτή τη στιγμή ε, εννέα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη Λιθουανία, αλλά τα τέσσερα από αυτά χρησιμοποιούνται από το 2000-2002, πάνω, εδώ και 10 χρόνια και πάνω δηλαδή, και δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, δεν αρκούν για τις ε, επιθεωρήσεις και τους ελέγχους μας. Ένα από τα ενδιαφέροντα εργαλεία που χρησιμοποιούν ε, τα τελωνία της Λουθωνίας είναι τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης των πινακίδων αυτοκινήτων και των ε, ε, κωδικών των εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποιούνται από το 2009 και ήδη έχουμε κατασχέσει τσιγάρα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ χάρη σε αυτό το σύστημα. Βλέπετε εδώ πώς λειτουργεί το σύστημα. Ε, έχει αναπτυχθεί και το σύστημα αυτό αναγνώρισης πινακίδων και κωδικών, ε, γιατί έτσι έχουμε την εικόνα της πινακίδας κάθε φορά. Ε, μπορούμε να εντοπίσουμε την άδεια λοιπόν κυκλοφορίας, την ταυτότητα του εμπόρευμα του κυβωτίου, ελέγχουμε στις μαύρες λίστες χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα και interface ή άλλες κινητές ε, συσκευές σε μόνιμη βάση. Και μπορείτε να δείτε το συντονισμό των δραστηριοτήτων μας, κοινή εκτίμηση κινδύνου, ανάλυση σε εθνικό επίπεδο. Το τελωνίο είναι η συντονιστική αρχή στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αγαθών. συμμετέχουν τέσσερις ε, αρχές, τα τελωνία, η αστυνομία, οι συνοριακές αρχές, αλλά και η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος. Έχουμε καθημερινές ε, αναφορές για τα διάφορα περιστατικά. και τα συστήματα μας χρησιμοποιούνται από το σε ε, αρχές ε, ε, αλλά και από την αστυνομία. Η συνεργασία τώρα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Ε, εδώ έχουμε μια ξεχωριστή πλατφόρμα βάση για την συνεργασία των τελωνιακών αρχών των βαλτικών χωρών. Ονομάζεται Via Baltica. Ε, οι επιχειρήσεις δηλαδή που κάνουμε. Υπάρχει ε, ένας δρόμος από τη Βαρσοβία αλλά και η Πράγα είναι υπό εξέταση γιατί η Τσεχία ζήτησε να μπει, ε, να συμμετέχει σε αυτές τις επιχειρήσεις. Η άλλη βάση που είναι μοναδική είναι η Task Force της Βαλτικής Θάλασσας για το οργανωμένο έγκλημα. Είναι μοναδική γιατί συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι της Ρωσίας εκεί. Και έχουμε τρεις οργανισμούς που αντιπροσωπεύονται εδώ είναι τα τελωνία, η αστυνομία αλλά και οι συνοριακές ε, αρχές. Ε, στις 4 ε, Απριλίου δε έγινε το τελευταίο βήμα σε αυτό το πρόγραμμα για αμοιβαία αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας ανάμεσα στις τρεις βαλτικές χώρες και αυτό μας επιτρέπει να ανταλλάσσουμε στοιχεία ε, online. Μπορούμε έτσι να στείλουμε προειδοποιήσεις, ε, να γίνουν ε, δηλαδή τελωνιακοί έλεγχοι σε άλλες χώρες και όπως είπα υπάρχει η συμφωνία, η νομική βάση για την ανταλλαγή στοιχείων ανάμεσα στις τρεις βαλτικές χώρες συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. Όπως βλέπετε, τα λιθουανικά τελωνία έχουν ε, επιτετραμένους στην Ένωση αλλά και στη Frontex αλλά και στην Ευρωπόλα, όπου γίνεται ο συντονισμός των ερευνών Υπάρχει συντονισμός από τον γύρο Τζαστή από τον Europol, όπως ίσως θα θυμάστε και από τα προηγούμενα παραδείγματα. Έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα συντονισμού από την Όλαφ. Κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, εμείς πιστεύουμε πως είναι οι ανθρώπινη πόροι, οι εξοπλισμοί, οι ε, λύσεις ε, της ε, τεχνολογίας, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς συνεργασίες και οικονομική πόροι. Υπάρχουν δύο είδη δραστηριότητας στο τελωνία στον αγώνα κατά της λιτουλάθρεμπορίου. Είναι η έλεγχη στα σύνορα και εντός της επικράτειας και η έρευνα, η εποπτεία και η επιχειρήσεις ε, μυστικές ε, επιχειρήσεις ε, για να αυξηθεί δε η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου χρειάζεται η αύξηση των εξοπλισμών και ε, ο εξυγχρονισμός τους, η βελτίωση της συνεργασίας των τελωνιακών αρχών ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης αλλά και με τις τρίτες χώρες, αλλά και η καταπολέμηση της διαφθοράς που είναι βασική για το τελωνίο μας, τα τελωνία μας πέρυσι και φέτος, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τα διοικητικά κόστη, την κάλυψη των διοικητικού κόστους. Και όπως ανέφερα στην αρχή της ε, παρουσίασής μου, τα κέρδη που προκύπτουν είναι η πιο επικίνδυνη ε, συνέπεια ε, γιατί επιτρέπει στο οργανωμένο έγκλημα να ε, ενισχύει τις δυνατότητες του να διαφθείρει, να υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρχές αλλά και στα δικαστικά συστήματα εν γέννη. Κάποιες ιδέες προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα είναι αφιερωμένο στην αγορά ελεκτικού εξοπλισμού για τα τελωνία, αλλά και ο καταμερισμός του κόστου συντήρησης. Υπάρχει σήμερα μεγάλη δυνατότητα, ε, μάλλον μια μεγάλη ποικιλία μέσων για την αγορά κινητών και σταθερών συστημάτων ε, ακτίνων Χ γίνεται υπό διάφορα συστήματα, πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ ελκυστικό, πρακτικό γιατί τα διάφορα προγράμματα διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και τα ποσοστά χρηματοδότησης και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες. Όπως, ε, όπως ίσως γνωρίζετε, είναι η ISA και η NPI, εξωτερικό, ε, μάλλον Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Και τέλος, θα πρέπει να, γίνονται να υπάρχει μάλλον συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τις εκστρατείες ενημέρωσης και κοινωνικής συνειδητοποίησης αλλά και ε, μη ανοχής για τα προϊόντα του λαθρεμπορίου και για τη χρήση αυτών από το κοινό. Το Ινστιτούτο Ελεύθερης Αγοράς της Λιθουανίας αναφέρει πως το 62% του πληθυσμού της Λιθουανίας δικαιολογεί τη χρήση των ε, ε, λαθρέων προϊόντων και το ίδιο το λαθρεμπόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Παϊγκοτζίνας. Το λόγο έχει ο κύριος Λάζεκ Παρδολομιέιτσικ. Oh, uh, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Thank Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά. Θα ήθελα να σας ε, μιλήσω από πλευράς ε, Πολωνίας σε σχέση με ε, την παράνομη εμπορία. Θα εστιάσω την προσοχή μου στην Πολωνία και μετά θα σας πω πώς μπορούμε γενικά να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο, ιδιαίτερα σε προϊόντα καπνού. Θα εστιάσω την προσοχή μου στα προϊόντα καπνού, διότι το παράνομο εμπόριο καπνού είναι βασικό πρόβλημα στα ανατολικά σύνορα, όπως, είπαν, όπως είπε και η Frontex και η Λιθουανία. Η Πολωνία είναι πολύ δύσκολο να, προσθέσει, να, συγγνώμη, να προστατεύσει τα εξωτερικά της ε, σύνορα, διότι έχει τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα, γιατί πρώτα έρχεται η Ουκρανία, η Λευκορωσία και μετά η Ρωσία. Επίσης ε, υπάρχει ε, το γεγονός ότι η Πολωνία είναι η ε, χώρα διέλευσης γιατί η Λευκορωσία και η Πολωνία μάλλον είναι πολύ ε, εύκολο από πλευράς Λευκορωσίας να γίνει διέλευση στην Πολωνία για το παράνομο εμπόριο. Επίσης, είμαστε πολύ επιτυχείς στην κατάσχεση τσιγάρων στα σύνορα βλέπετε ότι έχουμε πολύ καλές επιδόσεις, μιλάμε για 600 ε, δις. Ξέρουμε για ποιους λόγους γίνεται αυτό το παράνομο εμπόριο. Οι χώρες προέλευσης είναι η Λευκορωσία, η Ουκρανία και μετά η ε, ε, Ρωσία μέσω του θύλακα του Καλίνιγκρατ αλλά επέρχονται αλλαγές ως προς την ε, διέλευση. Όπως είπε και ο συνάδελφος από τη Λιθουανία, η Λιθουανία ήταν η βασική ε, χώρα διέλευσης. Αλλά από το 2010 έχει αλλάξει η κατάσταση και τώρα ε, η διέλευση γίνεται από την Λευκορωσία κατά ένα 60%. Και επίσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας νέος ε, διάβλος από τον Νότο, ο οποίος είναι αρκετά επικίνδυνος για την Πολωνία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τους ε, διάβλους υπάρχουν και θέματα τακτικής τα οποία είναι αρκετά ευέλικτα. Μέχρι λίγα χρόνια πριν γινόταν παράνομο εμπόριο ε, τσιγάρων, αλλά σε περιορισμένους διάβλους και μετά λόγω κατασχέσεων έχουν αλλάξει οι οδικοί αυτοί διάβλοι. Δηλαδή, πολύ συχνά βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση ε, των απολειών και πολλές φορές βλέπουμε ότι και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, πακέτα και λοιπά έχουν επέλθει αλλαγές. Άρα κυρίως από τη Λευκορωσία προέρχονται, ε, προέρχεται το παράνομο εμπόριο, αλλά και από τη Ρωσία και τη Μολδαβία. Όμως υπάρχει μία φθήνουσα πορεία, ενώ από τη Λευκορωσία έχει διπλασιαστεί το παράνομο εμπόριο. Δηλαδή μιλάμε για ένα 80% των αγαθών και γι' αυτό η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ε, μία συγκεκριμένη ε, στρατηγική και αυτό ισχύει και από πλευράς Λευκορωσίας γιατί, πολλές, ε, γιατί στο παρελθόν ο θύλακας του Καλίνιγκρατ ήταν ο μεγαλύτερος. Αλλά τώρα τα περισσότερα αγαθά προέρχονται από τη Λευκορωσία. Εδώ μιλάμε για παράνομα ε, αγαθά που δεν φέρουν ε, σήμα και που έχουν διεισδύσει στην αγορά. Ποια, ποιες είναι οι συνέπειες. Οι συνέπειες είναι πολύ σημαντικές Κάθε χρόνο χάνουμε 3,5 δις σλότης από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων. Δηλαδή μιλάμε για 8 δις ε, τσιγάρα που εισάγονται παράνομα στη χώρα. Μέσω μεγάλων κοντέινερ. Μιλάμε για ένα 10 με 12% του παράνομου εμπορίου. Υπάρχει ένα θέμα δημόσιας τάξης καταρχήν. Το παράνομο εμπόριο αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος στα σύνορα. Και το επίπεδο του παράνομου εμπορίου είναι της τάξης του 50%. Επίσης γίνεται επανεπένδυση κέρδους σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι τελωνιακές μας αρχές είναι ιδιαίτερα επιτυχείς στην κατάσχεση τσιγάρων. Δηλαδή η αρνητική τάση ε, έχει μετατραπεί σε θετική. Και από το 2009 βλέπουμε μία φθήνουσα πορεία του παράνομου εμπορίου αλλά όλα έχουν ένα αντίτιμο. Αν δείτε αυτό το γράφημα, βλέπετε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ευέλικτο, βρίσκει άλλους τρόπους διείσδησης και τώρα έχουν ε, επικεντρωθεί στο, στον κομμένο καπνό. Αυτό το βλέπουμε και στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Έχουν γίνει υψηλές, ε, πολύ μεγάλες κατασχέσεις. Υπάρχει μια νοδική πορεία και εδώ βλέπετε τις, ε, το επίπεδο των κατασχέσεων. Επίσης, έχουμε εκπονήσει μια στρατηγική καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου, ιδιαίτερα για τα καπνά και ιδιαίτερα από τη Λευκορωσία. Υπάρχει μία ε, task force που συντονίζει τις δραστηριότητες και υπάρχουν κινητές μονάδες σε όλα τα τελωνία, όπως βλέπετε σε αυτή τη γραφική παράσταση. Μιλάμε για πάνω από μισό εκατομμύριο κομμάτια παράνομου, παράνομου υλικού και όχι μόνο εντός Πολωνίας. και δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς ε, συνεργασία και ε, σε χώριο επίπεδο αλλά και διεθνώς. Δεν μιλάμε μόνο λοιπόν για προστασία των συνόρων, αλλά και για ε, συνεργασία προς τα έξω. Ένα μέρος, ένα τμήμα της στρατηγικής μας αφορά την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 73% των ε, πολιτών υποστηρίζουν το ενεχόμενο κόστος του καπνού εάν, υπάρχουν, εάν υπάρχει ένα μέρος δηλαδή χορηγείται για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Δηλαδή οι πολίτες δέχονται να αυξηθεί το κόστος των τσιγάρων για να αυξηθεί και η ασφάλεια. Τώρα πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Όπως βλέπετε το διεθνές εμπόριο έχει και διεθνή βάση γι' αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την παγκόσμια διάσταση του παράνομου εμπορίου. Υπάρχουν μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και το πιο συνεκτικό είναι η σύμβαση πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού και το πρωτόκολλο για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού. Και τις επόμενες ε, εβδομάδες θα έχουμε και την έγκριση της οδηγίας περί καπνών. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας των προϊόντων και αυτή είναι η καλύτερη λύση για να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο. Όπως σας είπα λοιπόν, έχουμε την σύμβαση πλαίσιο που εγκρίθηκε από 176 χώρες και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση της ε, προμήθειας, της, της ε, ζήτησης και της προσφοράς σε παράνομη, παράνομα είδη και φέτος, το 12 μάλλον, 140 χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν το σύστημα ανιχνευσιμότητας με βάση αυτό το πρωτόκολλο για την απαλυφή του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού. Προβλέπουμε λοιπόν ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας του παράνομου εμπορίου και προσπαθούμε να ελέγξουμε ε, τα τσιγάρα σε επίπεδο πακέτων Χρειάζονται πληροφορίες ε, για το, την αλυσίδα παραγωγής, το, την, ε, την χώρα όπου μεταβαίνουν και έχει σημασία να υπάρχει ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας το οποίο ε, δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ε, βιομηχανίας τσιγάρων. Αυτό είναι μέρος της τρέχουσας ε, πρωτοβουλίας. Και ο ζήτησε κάτι τέτοιο. Το σύστημα λοιπόν αυτό θα πρέπει να γίνει όλο ένα και πιο αποτελεσματικό. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, ε, καθώς και φυσική και ψηφιακή προστασία των αγαθών έτσι ώστε να έχουμε μία διαδικασία ταυτοποίησης, έλεγχο παραγωγής και έλεγχο διανομής. Επειδή αυτά τα, ε, τα συστήματα υπάρχουν σε αρκετές χώρες και σε μη ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούμε ότι για να υπάρχει ένα σωστό σύστημα ανιχνευσιμότητας, Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τεθούν στην εφαρμογή, δηλαδή θέμα ε, ε παγκόσμιου ελέγχου, ταυτοποίησης, ε, ελέγχου παραγωγής, διανομής κλπ. Μιλάμε λοιπόν για σήμανση των προϊόντων, σαφή συριακή ε, σήμανση όπως ισχύει και με τα χαρτονομίσματα. Δεν υπάρχει μόνο ένας ε, συριακός αριθμός και το αντίτιμο, αλλά ε, ορισμένα στοιχεία ασφαλείας ε, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει παραχάραξη. Το ίδιο θα θέλαμε να ισχύει και στην περίπτωση των σιγάρων. Επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε την αλυσίδα παραγωγής. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται από τη βιομηχανία καπνού, αλλά από τις κυβερνητικές αρχές, έτσι ώστε να γίνεται σήμανση σε κάθε προϊόν και να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πλήρης ανιχνευσιμότητα από τη σήμανση αυτή. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αφορούν όλες τις συσκευασίες από το πακέτο μέχρι την κούτα, μέχρι τις ε, συλλογικές συσκευασίες, τις μεγάλες συσκευασίες, έτσι ώστε να έχουμε ένα, μια σωστή ανιχνευσιμότητα. Το λεγόμενο σύστημα EMCS. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, πλήρη ανιχνευσιμότητα. Το ίδιο αφορά και τις επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιθεώρησης και αν υπάρχουν παραχαραγμένα προϊόντα θα πρέπει να καταγράφονται και οι πληροφορίες να αποσταλούν στο Υπουργείο έτσι ώστε να μην υπάρχει διαφθορά, να μην μπορεί δηλαδή να προωθηθεί η διαφθορά η εξαγορά. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στην ε, κυβέρνηση να ε, προβεί σε ίσπραξη φόρων, σε μεγαλύτερη ίσπραξη φόρων και με αυτή την ανιχνευσιμότητα η κυβέρνηση μπορεί να προβεί σε φόρο πολύ υψηλότερες. Και όταν αυξάνονται και οι φόροι, υπάρχει και κίνητρο για μεγαλύτερες ε, παραχαράξεις. Δηλαδή, αν δείτε όμως, ε, οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους φόρους, αλλά έχουν λιγότερες πράξεις. Με το σύστημα ανιχνευσιμότητας θα είμαστε σε θέση ε, να έχουμε περισσότερες εισπράξεις. Μιλάμε λοιπόν για την εφαρμογή αυτού του συστήματος και η εισπράξη σε μία χώρα ε, φόρων κατά 31% υψηλότερους στα καπνά. Και όταν, ακόμα και όταν αυξήθηκαν οι φόροι, και μειώθηκε ο όγκος παραγωγής, παρόλα αυτά εισπράττονται οι υψηλότεροι φόροι. Ως προς τις συστάσεις τώρα, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση την οδηγία περί καπνών, θα μπορέσουμε να πείσουμε τις ευρωπαϊκές ε, χώρες για την ε, ε, τάχιστη εφαρμογή του πρωτοκόλου FCTC και να ενθαρρύνουμε τις γείτονες χώρες να κάνουν το ίδιο. Γιατί και εμείς θα ευεργετηθούμε από κάτι τέτοιο. Έχει επίσης μεγάλη σημασία να ενσωματώσουμε ε, λύσεις που έχει ε, προτείνει και το πρωτόκολλο FCTC και να ενσωματωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Διαφορετικά θα υπάρχει κενό μεταξύ των δύο μηχανισμών. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα ανιχνευσιμότητας σε όλες τις ε, χώρες, ανεξάρτητα από τους ε, παραγωγούς. Επίσης να υπάρχει ασφαλή σήμανση των προϊόντων έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τους πολίτες μας. Να προστατεύσουμε δηλαδή και την δημόσια υγεία. Και τέλος, θα πρέπει να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των ε, τελωνιακών υπηρεσιών να υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα στα στοιχεία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ροζάλα. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούσαμε ήδη πως ε, από τους προλαλήσαντες πως τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται ε, επαρκώς και είναι επαρκώς εξοπλισμένα, οπότε θα εστιαστώ στην συνεργασία. Στα σύνορά μας Φιλανδίας με τη Ρωσία. Δηλαδή, πέρσι είχαμε γύρω στα 12 εκατομμύρια διελεύσεις. Αυτό σημαίνει πως γύρω στα 5 εκατομμύρια τουρίστες έφτασαν πέρσι στη Φιλανδία. Η πίεση λοιπόν στα σύνορα είναι τεράστια και η εσωτερική συνεργασία αστυνομίας τελωνίων και συνοριοφυλάκων ε, υπάρχει, ούτως ή άλλως υπάρχει στην νομοθεσία μας και θα επανέλθω σε αυτό. Τώρα πώς συνεργαζόμαστε στα σύνορα με τους ε, συναδέλφους μας της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχουμε συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε στα κοινά σύνορα. Έχουμε κοινά μέτρα. Έχουμε καλή ανταλλαγή πληροφοριών και τακτικές συναντήσεις και συζητήσεις με τις ε, ρωσικές αρχές. Ε, έχουμε μακρά ιστορία και η συνεργασία είναι καλή και καθόλου γραφειοκρατική. Συνεργαζόμαστε το υψηλό επίπεδο, στο κεντρικό επίπεδο και στο επίπεδο το επιτόπου. Τώρα, κάποια λίγα λόγια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε μία διπολική ε, αντιμετώπιση του ζητήματος. Έχουμε αφενός αστυνομία, τελωνία, συνοριοφυλακές και από την άλλη είναι η διοικητική διαδικασία επιλογής στόχων. Έχουμε λοιπόν τις πληροφορίες και την ανάλυση που γίνεται στα κέντρα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση και επιπλέον έχουμε και ένα κέντρο ανάλυσης ε, ένα κέντρο ανάλυσης όπως είπα που είναι το βασικό, ένα για τα λιμάνια, ένα για τα αεροδρόμια και ένα για την ξηρά. Η δομή είναι η εξής πρώτα απ' όλα. Τα κέντρα αυτά αστυνομίας τελωνίων και συνοριοφυλάκων συλλέγουν, να αναλύουν ε, τις ε, πληροφορίες και το προϊόν είναι μια αξιολόγηση κινδύνου και σχέδια δράσης. Βλέπετε πως σύμφωνα με τις επιχειρησιακές αναλύσεις μετά από αυτό μπορούμε να καθορίσουμε περιφερειακούς και εθνικούς ε, στόχους. Και άρα περνάμε μετά σε μια διοικητική διαδικασία επιλογής στόχων. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από την μονάδα έρευνων ή από κάποια μονάδα αστυνομία ε, τελωνίων συνοριοφυλακής. Καταγράφεται η απο καποια μοναδα αστυνομια τελωνιων φυλακης καταγραφεται η κινηση του στόχου, γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση από τα κέντρα αυτά και το αποτέλεσμα είναι ένας περιφερειακός ή εθνικός στόχος για, οργανω... για σοβαρό έγκλημα. Η συνεδρίαση για την επιλογή του στόχου είναι υπό την προεδρία του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης του Εγκλήματος, που ασχολείται με τη σοβαρή εγκληματικότητα. Μετά, όταν επιλεγεί ο στόχος, η αρμόδια μονάδα θα εστιάσει σε αυτόν και Ε, μετά η αρμόδια αυτή μονάδα ενισχύεται με επιπλέον πόρους. Και τέλος, το τελευταίο σημείο αφορά την, ε, το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα στη και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες. Μιλάμε όχι μόνο για ρωσικό οργανωμένο έγκλημα, αλλά για ρωσόφωνο οργανωμένο έγκλημα. Η Φιλανδία και άλλες χώρες ε, επηρεάζονται εμέσως. καθώς είναι προμηθευτές της σκιώδους οικονομίας και συνδέονται μέσω διαφόρων εταιριών. Το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα σημαντικό τομέας εγκληματικότητας ε, και εδώ πέρα έχουμε δραστηριοποίηση του ρωσόφωνου εγκλήματος και θεωρείται πως και κάποιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων ξεπλένουν χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες. Η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη απειλή και Έχουμε ε, άρα ζητήματα που αφορούν και τα τελωνία, όπως τα διπλά τιμολόγια και τέτοια πράγματα, λαθρεμπόριο και τέτοια πράγματα. Καθώς λοιπόν πάρα πολλές εταιρείες ε, επιμελητίας και φοδιασμού μεταφορών είναι στα χέρια Ρώσων, υπάρχει αρκετά μεγάλη σύνδεση με το έγκλημα. Συχνά η Ρωσική Ομοσπονδία είναι επίσης χώρα από την οποία προέρχεται ηλεκτρονικό έγκλημα και εκεί πέρα καταλήγουν και τα έσοδα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ξαφρίσματος των στοιχείων πιστοτικών καρτών και είχαμε πολλές αποκαλύψεις τέτοιων στοιχείων. Τι γίνεται τώρα με τα ναρκωτικά. Ήδη αγορά η ηρωίνη στη Ρωσία και η Ουκρανία είναι μεγαλύτερη από την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια ηρωίνη μπαίνει στη Ρωσική Ομοσπονδία από Λιθουανία και Λετωνία αλλά και από άλλες χώρες. Και υπάρχουν επίσης και συνθετικά ναρκωτικά και η κοκαίνη η οποία ενισχύεται και προϊόντα αμφεταμίνης ειδικά στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης και της Φιλανδίας. Επίσης, η Φιλανδία είναι μια χώρα διαμετακόμισης για κοκαίνη και ρητίνη κάναβης που πάει προς την Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και άλλα ναρκωτικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κυρίε και κύριοι. Σας ευχαριστώ. Για τη συζήτηση θα αφήσω το Προεδρία στον κύριο Κύρκοπ. Ladies um, Κυρίες και κύριοι, να η ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις στους ομιλητές, καθώς και να σχολιάσετε τα όσα ακούσατε. Πρώτος σας το κατάλογο είναι ο κύριος Γιακολίνο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις τέσσερις διαδοχικές ε, παρεμβάσεις που ενίσχυσαν την πεποίθησή μας ε, που μπορεί και από το περιεχόμενο των ε, όσων έχουμε ήδη συζητήσει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, στις δικαστικές αλλά και στις τελωνιακές εκεί που χρειάζεται ανάμεσα στις χώρες μέλη αλλά και με τρίτες χώρες για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ε, όλα τα εγκληματικά φαινόμενα, κυρίω αυτό που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Πρώτη μου ερώτηση αφορά τον κύριο του διευθυντή Ρόσλαρ του Frontex. Έχουμε προβλέψει τη δημιουργία μιας υπηρεσίας στο εσωτερικό του Frontex ακριβώς για να ενισχυθούν οι δραστηριότητες ε, κατά του λαθρεμπορίου, του εμπορίου ανθρώπων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Μιας υπηρεσίας που θα μπορέσει να παρακολουθεί καλύτερα τις ε, δραστηριότητες μας ακριβώς Πρόκειται για μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ακτοφυλακής. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τη γνώμη σας, τη γνώμη της Frontex σε σχέση με τη δημιουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας που θα συζητήσω και με τους υπόλοιπους συναδέλφους και τους κυρίως τους σκιώδες. Τώρα από τον ε, υπεύθυνο των ε, τελωνιακών αρχών της Λεφανίας αλλά και τους αντίστοιχους της Πολωνίας και της Φιλανδίας προέκυψε από τις παρεμβάσεις σας η βασική ανάγκη για παράδειγμα του Διευθυντή Τελωνιακών Αρχών, αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων που καλύτερα θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις εγκληματικές ενέργειες και μέσω της συνεργασίας με την Ιντερπολ, επίσης επισήμαση προϊόντων για να αποφύγουμε υποθέσεις ε, παραχάραξης ή πλαστών ε, προϊόντων, το θέμα της αντίθεσης της διαφθοράς με την ανακύκλωση, συστήματα που μπορούμε να ε, νικήσουμε μόνο αν διαφερηθούν τα σύνορα στις επικράτειες των κρατών μελών. άρα λοιπόν και οι δικές μου σκέψεις επιβεβαιώνονται και επιβεβαιώνονται και από τις δικές σας παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Anyone else like to raise any questions at this point? Um... Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι αυτή τη στιγμή. Σμιτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άργησα λίγο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά άκουσα τον Φιλανδό κύριο. Εγώ είμαι από τη Σουηδία και ανησυχώ ιδιαίτερα για τη ρωσική μαφία που έρχεται στις σκανδιναβικές χώρες. Και είπατε πως πολλά από αυτά, πολλές από αυτές τις δραστηριότητες διέρχονται από τη Φιλανδία και υπήρχαν πολλές κατηγορίες πως το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα έχει εγκατασταθεί στις χώρες μας. Και το ερώτημά μου είναι πώς πρέπει να αντιδράσουμε. βοηθάνε καθόλου οι Ρώσοι. Ο κύριος Πούτιν κάνει τίποτα. Εγώ θεωρώ πως μάλλον το αντίθετο κάνει. Αλλά ίσως μπορείτε και εσείς να μας εξηγήσετε. Κοιτάξτε. Όσο σκέφτονται οι υπόλοιποι, νομίζω καλό είναι να ζητήσω από το πάνελ να απαντήσει σε ερωτήσει. Ναι, Κύριε Ρέσλερ, ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω πως δεν είμαι ακριβώ σίγουρος για το να κατάλαβα τι εννοείται. αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ιακολίνο. Η Frontex, λόγω της εντολής της, εστιάζει στην βελτίωση του ελέγχου των συνόρων και όταν λέμε έλεγχο συνόρων μιλάμε για την αποτελεσματική καταπολέμηση του διασυνοριακού σοβαρού εγκλήματος. Και άρα στόχος είναι μαζί με τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα να απτύξουμε τις κοινέ μας επιχειρήσεις για να καταλήξουμε σε κοινέ επιχειρήσει με πολλαπλούς στόχους. Και προσπαθούμε να βελτιώσουμε βεβαίως τη συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και χωρών για να μπορέσουμε να εγκνεύσουμε την παράνομη μετανάστευση και άλλα είδη διασυνοριακού εγκλήματος, παραδείγματος χάρη στη θάλασσα. Τα σκάφη μεταφέρουν ναρκωτικά, ας πούμε, από τη Βόρεια Αφρική στην Ισπανία. Δεύτερον, έχουμε στόχο να ενισχύσουμε τον τοπικό έλεγχο στα συνοριακά φυλάκια. Αυτό μπορεί να γίνει, όπως είπα, μέσω των σημείων εστίασης, στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεργασία τελωνιακή που είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα υποστηρίζεται κυρίως στο εθνικό επίπεδο και με την ομάδα εργασίας τελωνίων και με τη συνεργασία μέσω του Όλαφ. Και υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την συνεργασία μέσω της τοπικής, τοπικού συντονισμού, π.χ. στη Βαλτική, όπου έχουμε την πολύ γνωστή συνοριακή συνεργασία της Βαλτικής. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει η Frontex από την εντολή της, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω πως πρέπει να σκεφτούμε και τους περιορισμούς της εντολής μας. όσον αφορά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. κύριος Παγκασίνης. Μάλιστα. Το βασικό ερώτημα αφορούσε την τελωνιακή συνεργασία. Και ποια υπηρεσία μπορούσε να συντονίσει. Ο συνάδελφος ανέφερε την ομάδα συνεργασίας των τελωνίων που είναι αρμόδια για αυτές τις επιχειρήσεις και αφορά βεβαίω και τις τελωνιακές ε, δραστηριότητες όσον αφορά τη συνεργασία με τις υπηρεσίες συνοριοφυλακής η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλύτερη ε, πιο δομημένη θα έλεγα Και, ως έναν βαθμό. Νομίζω πως επιτύχαμε το βασικό μας στόχο. Και βεβαίως πάντα υπάρχει νομίζω περιθώριο βελτίωσης, αλλά νομίζω πως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Κύριος Μπάρτλερ. Ευχαριστώ. Για να προσθέσω κάτι ακόμα. Θεωρώ πως, όπως είπα, είναι ένα πράγμα η προστασία των συνόρων και όλες οι υπηρεσίες, τελωνία κτλ. πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγουν οι κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. και στα δικά μας κατημέλη και σε άλλες χώρες θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία, όπως είπα, της ε, διεθνούς ε, συνεργασίας και φορέων όπως η FCTC. Υπό την αιγίδα τέτοιων ε, οργανισμών, εάν εφαρμοστούν όλες οι στάσεις, όλες οι υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για διακίνηση παρανόμων αγαθών και ε, θα είναι ορατή η διακίνησή τους. Ένας τρόπος καταπολέμησης είναι αυτός. Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλα τα παράνομα αγαθά, τα λαθρέα, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Σε ό,τι έχουμε, ε, βεβαίως ανταποκρινόμαστε. Η βάση δεδομένων ε, είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Νομίζω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για τη ρωσική μαφία, θα πρέπει να μιλάμε για το ρωσόφωνο οργανωμένο έγκλημα. Δεν πρόκειται μόνο από, για τη Ρωσία, αλλά από, τις, ε, από την ε, κοινοπολιτεία γενικότερα. θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο εκκίνησης, δηλαδή συνεργασία με τρίτες χώρες, μιλώντας και για τη Ρωσική Ομοσπονδία. Χρειάζεται, χρειάζονται πρωτόκολλα, προγράμματα δράσης, συνεργασία, συμφωνίες. Θα πρέπει να ορίσουμε κοινούς στόχους και κοινή δράση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Σε επίπεδο Σκανδιναβίας και βορείων χωρών έχουμε μία μακρά παραδοσιακή συνεργασία και υπάρχει και ένας ειδικός φορέας συνεργασίας των αστυνομικών αρχών. Άρα ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές που διαθέτουμε για να ασχοληθούμε με το ρωσόφωνο έγκλημα. Και αυτό αφορά και τη Βαλτική μέσω της Task Force που σας προανέφερα. Ευχαριστώ. Κύριε Λένε, Είπατε ότι έχετε μία συμπληρωματική ερώτηση και μετά ο κύριος Νιούτον Ντάν μπορεί να υποβάλει τις ερωτήσεις του. Ο κύριος Γιακολίνο, ίσως δεν ήμουνα σαφής ως προς την ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Frontex. Η ερώτηση είναι εξής. Οι αρμοδιότητες της Frontex είναι γνωστές. Το Μάρτιο του 2011 στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έγινε λόγος για αυτές τις αρμοδιότητες. Στην πρόταση του εισηγητή γίνεται λόγος για το εξής για τη δημιουργία μιας ε, ακτοφυλακής που θα ήταν ένας φορέας μέσα στη Frontex για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο από παραχάραξη, ναρκωτικά, οριοθετώντας και ελέγχοντας τα εσωτερικά και εξωτερικά θαλάσσια σύνορα. Το βλέπετε αυτό σαν υπόθεση εργασίας. Ποια είναι η θέση της Frontex. Και αν μπορεί να μας απαντήσει ο εκπρόσωπος της Frontex αλλά και η τα άλλα μέλη του ε, πάνελ. Κύριε Ρέσλερ, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε τώρα ή στη συνέχεια, συνοψίζοντας, αν θέλετε μπορείτε και τώρα να απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί βασική αρμοδιότητα και μέλημά μας. Και υπάρχουν και οι αρχές για τον έλεγχο των συνόρων μέσω ακτοφυλακής. Αυτό είναι αναπόσπαστο στοιχείο των αρμοδιοτήτων μας. Άρα η Frontex δεν μπορεί να προωθήσει το θέμα της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής. Αυτό εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη εδώ και δύο-τρία χρόνια ασχολούνται με θέματα ακτοφυλακής έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή που να υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη και η Frontex. αλλά εναπόκειται στα κράτη-μέλη να την ορίσουν, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά θαλάσσια ασφάλεια και άλλες αρμοδιότητες. Πρόκειται για πολλές εμπλεκόμενες αρχές. Μιλάμε για εφαρμογή ε, του, ε, του δικαίου και κυρίως του αστικού. Αυτή είναι η θέση της Frontex επί του θέματος. Ευχαριστούμε. Νιούτον Ντάν. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε. Ψήφιζα σε μια άλλη επιτροπή. Ε, δεν είδα τις παρουσιάσεις σας. Ελπίζω να μας αφήσετε το υλικό. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία προς τον κύριο Ραγιάλα. Δεν θεωρώ πως απαντήσατε στο ερώτημα του κυρίου Σμίτιν. Ο Πούτιν είναι μαζί μας ή εναντίον μας βοηθάει ή δεν βοηθάει. Α, θα θέλαμε να το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, αν θέλετε να απαντήσετε, καταλαβαίνω. Ε, και αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό. Για τους κυρίους δε που μίλησαν, μπορείτε να μας πείτε ένα πράγμα που θα θέλατε να αλλάξει. Αυτή η δουλειά της ε, Επιτροπής μας για να σας βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Τι θα θέλατε λοιπόν να μας προτείνετε. Ναι, νομίζω πως θα ακούσουμε όλους τους ομιλητές, νομίζω πως ε, είχα ασχοληθεί βεβαίως με τα ζητήματα πουτινολογίας πριν από λίγα χρόνια. Αν έχετε κάποιες πληροφορίες, ευχαρίστω. Τώρα δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη σημερινή μας συζήτηση. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Παραζίνης. Πάγελα, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Ας ξεκινήσουμε από εσάς και μετά στον κύριο Ράγκλη. Είναι δύσκολο να επισημάνω ένα ζήτημα, αλλά αν επιμένετε θα έλεγα, την ευαισθητοποίηση. Όσον, για να μην, ε, γίνεται, να μην γίνονται ανοιχτά τα λαθρέα προϊόντα. Γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες, τα εγκλήματα δηλαδή, κατασχέσεις προϊόντων, αλλά ο στόχος είναι να αλλάξει η νοοτροπία, να πέσει η κατανάλωση, η ζήτηση. Αυτός είναι ο στόχος. Α, ο κύριος Ραγιάλα. Τώρα δεν ξέρω για τον κύριο Πούτιν. Ε, ίσως δεν είμαι και ο κατάλληλος άνθρωπος για να θέσω εγώ το ερώτημα στον κύριο Πούτιν. Ίσως στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα μπορούσε κάποιο να το θέσει. Τώρα για το θέμα της συνεργασίας. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας. Για το θέμα του αυτό υπάρχει και μια ομάδα εργασίας που επισκέφθηκε τη Μόσχα και αφορούσε τις ε, θεωρήσεις των διαβατηρίων. Ήταν οι περισσότερες διοκτικές αρχές εκεί πέρα και συζητήσαμε την εγκληματικότητα και τη συνεργασία και πάντα υπάρχει όπως είπα, περιθώριο βελτίωσης της συνεργασίας, αλλά το βασικό μήνυμα ήταν πως τα Υπουργεία που είναι αρμόδια και οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας συνεργάζονται. Και είναι και πολύ ειλικρινείς και πολύ ανοιχτές. Κάποιος άλλος θα ήθελε να σχολιάσει κάτι. Ναι, παρακαλώ. Για το ερώτημά σας, για τις συστάσεις. Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε τη ζωή δύσκολη σε λαθρεμπόρους και λοιπούς. Αυτό με έναν τρόπο μπορεί να γίνει. Το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία Ε, για να εμποδιστεί, όπως είπα, η παραγωγή και να κερδίσουν και περισσότερα χρήματα τα κράτη, έτσι. Ανέφερα το παράδειγμα του καπνού. Πήχε να υπάρξει ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης ε, των ε, λαθρέων αγαθών. Εάν δηλαδή με ασφαλή τρόπο σημαδεύεται και σημαίνεται η νόμιμη παραγωγή, θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη ε, η δραστηριοποίηση των ε, λαθρεμπόρων. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω θα ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Μάλιστα, κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι. Μάλιστα. Τότε θέλω να σας ευχαριστήσω. για τη συνεισφορά σας και η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 7 Μαΐου και νομίζω θα ψηφίσουμε μια διάμεση έκθεση. Αυτή είναι η επόμενη συνεδρίασή μας λοιπόν. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.